Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω στην απόγευματινή συνεδρίαση της ΣΥΜΚΟ. Περνάμε με το, στο σημείο 9, την έκθεση δηλαδή για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Η συγκητής μας είναι ο Παύλο Αρίας Ετσεβερία. Ελπίζω να μην κατακρεωρίσω το επίθετό σας κύριε Ετσεβερία από το ΕΛΚ. Θα ήθελα πρώτα σας να δώσω το λόγο, μετά στους και οδησίγητες και στα υπόλοιπα μέλη της ΣΥΜΚΟ και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο κύριε Τσεβερία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας καταρχήν. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ε, σκιώδης ηγητές για την πολύ καρποφόρα συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις τροπολογίες και τους ευχαριστώ και για τις ε, συμβαστικές τροπολογίες που ομαδοποίησαν τις πολύ χρήσιμες και εύστοχες τροπολογίες των συναδέλφων. Είμαι γενικώ ικανοποιημένο και από το αποτέλεσμα, αλλά και από τις συμβαστικές λύσεις ε, που βρήκαμε χάρη στη συνεργασία των πολιτικών ομάδων. 110 τροπολογίες συνολικά υποβλήθηκαν και Καταλήξαμε σε 8 συμβαστικές τροπολογίες για πολύ σημαντικά θέματα, όπως το 5 για τις ε, υπηρεσίες αποστολής, για το ΦΠΑ, το 6, ε, πνευματικά δικαιώματα, 7 και προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, συμβαστική λύση 8. Όπω είπα και στο παρελθόν, η ολοκλήρωση τη ενιαία ψηφιακή αγορά αποτελεί ζωτικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που καλό θα ήταν να υλοποιηθεί στη διάρκεια τη δική μα κοινοβουλευτική θητεία. Χαίρομαι ιδιαίτερω λοιπόν που σε γενικέ γραμμέ όλε οι πολιτικέ ομάδε συμφωνούν με αυτό το στόχο της ανάγκης ολοκλήρωση τη ενιαία ε, ψηφιακή αγορά, όπω φάνηκε και από την ε, ομόνια που επικράτησε στι ε, συναντήσει που είχαμε τους σκιώδει ηγητέ. Όπω όλοι ξέρουμε, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα ανέλαβαν τα τελευταία δύο χρόνια πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για να αντιστραφεί η παρούσα κατάσταση και να υπερκεραστούν οι φραγμοί που ακόμη και σήμερα μας εμποδίζουν από την αξιοποίηση των πραγματικών πλεονεκτημάτων μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στην Επιτροπή μας εγκρίναμε πολλές εκθέσεις και νομοθετικά ψηφίσματα όπως το 2010 για την ολοκλήρωση Τη ε, αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή, την έκθεση για την ε, ενιαία πράξη της ε, εσωτερικής αγοράς για τους Ευρωπαίους, τον κανονισμό για τα εναλλακτικά συστήματα επίλυση διαφορών και πολύ σύντομα θα εγκρίνουμε και τον κανονισμό για την ηλεκτρονική υπογραφή. Επίσης είχαμε και την ομάδα εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ψηφιακή αγορά. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί η υποστήριξη της Επιτροπής για τη συνέχιση των εργασιών προκειμένου να κρατήσουμε ένα ανοιχτό φόρουμ ε, συζητήσεων και προβληματισμού που θα μας βοηθήσει και στη συνέχεια των εργασιών μας. Τις επόμενες μέρες θα υποβληθεί στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων μια νέα πρόταση για το πρόγραμμα της ομάδας εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έχει εκδώσει διάφορες ανακοινώσεις και νομοθετικές προτάσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση της ενίας ψηφιακής αγοράς. Μεγάλη σημασία από αυτή την άποψη είχε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εμπόριο του Ιανουαρίου του 2011. Η ανακοίνωση αυτή προβλέπει ένα μεγάλο φάσμα προτάσεων και έναν οδικό χάρτη για την υλοποίησή τους, ε, θεωρώντας την ε, ολοκλήρωση της ε, ενιαίας ψηφιακής αγοράς την απαραίτητη διάσταση του Single Market Act 2 που υπευλήθη την περασμένη εβδομάδα. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε δύο θεωρώντας και μια αιτιολογική σχέση και σε μια προφορική τροπολογία που έστειλα στους και οδησηγητές και πριν από λίγο έδωσα και στα μέλη ε, της Επιτροπής, ενώ στη διάρκεια της απογευματινής συνεδρίας θα σας στείλω και τον ενημερωμένο κατάλογο ψηφοφορίας. Άμα επιτρέπετε θα ήθελα να σας διαβάσω πρώτα την προφορική τροπολογία που προτείνω. Θα τη διαβάσω λοιπόν, ε, θεωρώντας ένα. Λαμβάνοντα υπόψη την ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη 3η Οκτωβρίου του 2012, ανακοίνωση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο ε, Δεύτερη πράξη για την ενιαία αγορά, Single Market Act 2, Λέει λοιπόν η προφορική τροπολογία, καλωσορίζει τη νέα ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δεύτερη εκδοχή τη πράξη για την Ευρωπαϊκή Αγορά που περιλαμβάνει ε, σημαντικές δράσεις για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας. Ε, υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρου ε, αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων τη ψηφιακή αγορά. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ε, προφορική τροπολογία. Με την έκθεση αυτή προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη και τις εργασίες της ομάδας εργασίας για την ψηφιακή αγορά και θέλουμε να συμπληρώσουμε και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία που έχει η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να εισέλθουν και να εξοποιήσουν την ψηφιακή αγορά για να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση και να αναπτυχθούν οικονομικά. Αυτά προς το παρόν. Με ενδιαφέρουν πρώτα απ' όλα οι απόψει των σκιωδών εισηγητών αλλά και των υπόλοιπων μελών της, Ευρω... της Επιτροπής μας και ευελπιστώ ότι θα τύχω της υποστήριξη των πολιτικών ομάδων για την έκθεσή μου προκειμένου να συνεχίσουμε την καλή μας πορεία στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Ευχαριστώ. Thank you, Antonio, thank you for Ευχαριστώ, Αντώνιο, και ευχαριστούμε θερμά για το έργο σου σε αυτό το πολύ σημαντικό ντοσχέ που αποτελεί το αντικείμενο της έκθεσής σου. Τώρα από τους και οδησηγητές ο Αντώνιο δυστυχώς έμεινε στο Κιώτο λίγο παραπάνω θα έρθει αργότερα το απόγευμα θα ήθελα να υποβάλω τέσσερα σχόλια εκ Αντώνιο. Καταρχήν, οι συμβαστικέ τροπολογίε αποτελούν τον καρπό τη ε, επικοδομητική συνεργασία με τον κύριο Αρία και ανταποκρίνονται στην ανάγκη για μια διαφανή ε, και ρυθμισμένη ψηφιακή, ενιαία ψηφιακή αγορά που θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για μια ευφυή ε, οικονομική ανάπτυξη που δεν θα αποκλείει κανέναν. Θεωρούμε ότι η υλοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου για όλες τις ε, πτυχές της ε, ενιαίας αγοράς ε, θα πρέπει να αποφεύγει κατακαιρματισμό στην ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλίσουμε αυστηρότερους ελέγχους των κοινωτικών θεσμικών οργάνων ό,τι αφορά την σωστή εσωμάτωση της οδηγίας αυτής στην Εθνική Ένωμη Τάξη. Γιατί ο κατακαιρματισμός μέχρι στιγμής οφείλεται, οφείλεται είτε στην καθυστερημένη είτε στην προβληματική εσωμάτωση. Σε ό,τι αφορά τις ε, τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, είναι σημαντικό να προβλέψουμε και νέες ευρηματικές μορφές παράδοσης και να αναλάβουμε μέτρα που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και την απομόνωση των απομακρυσμένων περιοχών. Μια ενιαία ψηφιακή αγορά θα επιτρέψει στους καταναλωτές ε, ε, ένα μεγαλύτερο φάσμα επιλογών σε πιο ανταγωνιστικές τιμές και τέτοια δυνατότητα θα πρέπει να την έχουν όλοι οι καταναλωτές χωρίς καμία εξαίρεση. Ακόμη και οι καταναλωτές που διαμένουν σε περιφερειακές ε, ε, ζώνες ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο Αντώνιο Κορέα Δεκάμπος είναι πεπισμένος ότι το κείμενο της έκθεσης που θα ψηφιστεί αύριο θα αποτελέσει σημαντικό ρόλο στο νομοθετικό έργο των επόμενων ημερών που θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από τους φιλελευθέρους, ο κύριος Μπεζόη. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Εξ ονόματος του κυρίου Λόκεγκαρντ μου ζήτησε να πάρω το λόγο. γιατί δεν μπορούσε να είναι εδώ ανάμεσά μας. Η ψηφιακή ατζέντα εισαγωγικά είναι κάτι το κομβικό για την φιλελεύθερη ομάδα και μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να βγει από την κρίση. Θεωρεί ο κ. Λόκεργκάρντ ότι ο εισηγητής προσπαθεί έχει κάνει καλές προτάσεις και μέσω των συμβιβαστικών τροπολογιών. Έχει φέρει στην επιφάνεια τα προβλήματα της ψηφιακής αγοράς, διαφορά τιμολόγησης των ιδίων προϊόντων online και ε, εκτός ηλεκτρονικού εμπορίου, πολυδιάσπαση της αγοράς, θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεργασία και θα υποστηρίξουμε πάντα τον εισηγητή. Ο κ. Σένστρομ από τους Πρασίνους. Θα συμφωνήσω με τον εισηγητή και με τους προηγούμενους ομιλητές για τη σημασία της ηλεκτρονικής αγοράς αλλά και τις δυσκολίες που παρουσιάζει Είναι αλήθεια ότι απαιτούνται νομοθετικές ενέργειες για να πετύχουμε την επίλυση των προβλημάτων. Δεν συμφωνώ με τη συμβιβαστική όμως παρήθμη 7. Μια οδηγία για την επιβολή δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστέψει κανείς ότι μια αυστηρότερη επιβολή της προστασίας των προστασίας του, του δημιουργού μέσω των πνευματικών δικαιωμάτων είναι κάτι το πάρα πολύ περίπλοκο και αυτό πρέπει να επιδιώξουμε αν πράγματι θέλουμε εμείς να βρούμε νομικές επιπλέον ρυθμίσεις στην Ευρώπη, ε, ίσως θα πρέπει να καταστήσουμε ε, ικανές επιχειρήσεις όπως το Spotify να δώσουν πανευρωπαϊκές λύσεις. Πάντως η συμβιβαστική πρόταση ως έχει είναι προβληματική γιατί υψώνει πάρα πολλά εμπόδια στους ε, συμμετέχοντες στην αγορά αυτή. Δεν μπορώ λοιπόν, αστυνόμευση ε, σε εισαγωγικά επιπλέον δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Μακλάρκιν από τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ τον κύριο Αρία Σετσεβερία για την εξαιρετική δουλειά. Τον ευχαριστώ και για τις συμβιβαστικές τροπολογίες θα ήθελα να τον στηρίξω στις προτάσεις τις οποίες κάνει για την επιμόρφωση των εμπορευομένων online, την κατάρτιση μάλλον. Έχουμε καταθέσει πολλές τροπολογίες που υποστηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη συμμετοχή τους στο ευρύ φάσμα online, και προσπαθούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε καλύτερα την οδηγία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των καταναλωτών, συγγνώμη. Για την συμβιβαστική 7 δεν είμαι κατά της οδηγίας επιβολής, εγώ είμαι υπέρ αντίθετα, αλλά νομίζω ότι καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω εναλλακτικές λύσεις, διαφορετικά πρότυπα, έτσι ώστε να δούμε τι θα γίνει με το, με το φαινόμενο του licensing, της αδειοδότησης. Έχω καταθέσει λοιπόν αρκετές τοπολογίες, ελπίζω αυτές να γίνουν δεκτές από την Επιτροπή και να στηριχθούν από τον εισηγητή. Συγχαρητήρια λοιπόν για την εξαιρετική σας προσπάθεια. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα ήθελε το λόγο από την ΚΟΕ. Θα στραφώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω ποιος από σας τους δύο θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής για τα σχόλια τα οποία κάνατε. Δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε σε αυτά τα οποία ήδη είπατε και τις προηγούμενες εβδομάδες είπαμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε για την δουλειά που έχετε κάνει. Είμαστε ευγνώμονες προς τον κύριο Ετσεβερία. Τώρα από εδώ και πέρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα βάλουμε σε εφαρμογή όλα αυτά. Ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες να ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση Δεν θα μείνουμε στη διαβούλευση. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας και ένα οδικό χάρτη για να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς που μας αφορά. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν αναφέρεται εδώ αλλά νομίζω παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι πριν από το τέλος του μήνα θα υιοθετήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης και για τα ε, παίγνια online Νομίζω ότι αυτό έχει συζητηθεί ε, εκτενώς ε, τον προηγούμενο χρόνο. Τώρα πλέον κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Μετά ε, υπάρχει επίσης το θέμα των υπηρεσιών πληρωμών. Κρίσιμο για το σύστημα, κρίσιμο για τις εμπορικές δραστηριότητες και για τους καταναλωτές που δεν θα πρέπει να τους κοστίζει πάρα πολύ η διαδικασία αυτά. Αυτή. Έχουμε ξεκινήσει τη διαβούλευση για τα συστήματα πληρωμών. Τώρα περιμένουμε ε, την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών, η οποία θα έρθει του χρόνου. Θα υπάρξει επίσης ε, και το θέμα των ε, δαπανών που απαιτούνται για ανταλλαγή χρεώσεων με πιστοτικές κάρτες. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε από το πρόγραμμα δράσης πλέον σε πρακτική εφαρμογή και να καταστήσουμε την ηλεκτρονική αγορά να λειτουργεί ορθότερα και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και για την καλή σας δουλειά. Ελπίζω να προχωρήσουμε με ταχύτητα. Κλείνει λοιπόν το θέμα αυτό. Περνάμε τώρα στο σημείο 10 για την οδηγία που το, τα προτάσεις που τροπολογούν την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα. Η κυρία Βερνιό έπρεπε να είναι παρούσα κανονικά, αλλά δεν έχει έρθει ακόμη. Για να δούμε καταρχήν ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ή μήπως να αναλάβουμε, αναβάλουμε, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να δούμε πότε θα έρθει η κυρία να δουμε ποτε θα ερθει η κυρια βερνιό. Uh, now when we have the uh, time and uh, our beloved chair uh, Malcolm has already uh, arrived. Έχει επιστρέψει ο φίλτατος πρόεδρος Malcolm Harbour Πείτε μας λίγα λόγια για το πρόγραμμα. Ευχαριστώ και σε ευχαριστώ που προέδραψες στην απογευματινή συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η επόμενη εβδομάδα είναι και επισήμως η εβδομάδα εορτασμού των επιτευγμάτων της ε, ενιαίας αγοράς. Ε, και η αρχική έκθεση του, για την ενιαία αγορά υποβληθηκε το 1995. Συνάντησα χθες μια Βρετανίδα συντηρητική που το 98 υπέβαλε την έκθεση εκείνη και μου είπε ότι είχαν υποβληθεί 287 προτάσεις στο αρχικό πρόγραμμα για την εσωτερική, για την ενιαία αγορά. Βλέπετε ότι τώρα έχουμε πια μόνο 12. Έχουμε σημειώσει αρκετή πρόοδο. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και στο θέμα τη ολοκλήρωση τη ψηφιακή αγορα. Πάντω, τη Δευτέρα από τι 9 το πρωί, αν δεν κάνω λάθο ή 9.30, δεν θυμάμαι καλά. Α, 10. Εν πάση περιπτώσει, Δευτέρα το πρωί. Κάποια στιγμή θα έχουμε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η αρμόδια τη ομάδα μα τη Επιτροπή για τη σχέση με τον τύπο, είπε ότι με ενημερώνει ότι βρίσκονται online οι πληροφορίε και το όλο πακέτο. Ε, οπότε μπορείτε να επωφεληθείτε από την ενημέρωση αυτή για να εκδώσετε και σε ανακοινωθέντα τύπου για τα επιτεύγματα της εσωτερικής αγοράς. Η διάσκεψη αυτή λοιπόν θα λάβει χώρα τη Δευτέρα. Τα εγγένειά της θα γίνουν από τον πρόεδρο Μπαρόζο και τον υποφαινόμενο, γιατί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Σούλτς, θα πάει στο Βερολίνο. 9 10 λοιπόν το πρωί της Δευτέρας θα πρέπει να με ξαναϋποστείτε στα εγγένεια αυτή τη διάσκεψης. Ευελπιστούμε ότι θα δώσει το παρόν και ο πρώην πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ζακ Τελόρ. Τον περιμένουμε. Και από ό,τι ξέρω, θα απευθύνει μήνυμα μέσω βίντεο και ο κύριος Μόντι. Θα συμμετέχουν ε, κορυφαία μέλη της Επιτροπής, ε, Γκέρεκ, Σβάπ, κυρία Τιούν, ο κύριος Μάντερς, Ή, αυτοί είναι όλοι. Όλα αυτά τα σημαντικά θα γίνουν Δευτέρα πρωί. Ελπίζω να δώσετε και άλλοι το παρόν να είναι σημαντική αυτή η εναρκτήρια διάσκεψη. Φαντάζομαι θα έχετε λάβει προσκλήσεις και για αντίστοιχε εκδηλώσεις στις πατρίδες σας. Την πέμπτη το απόγευμα εγώ θα μεταβώ σε αντίστοιχη διάσκεψη στο Λονδίνο. Και όσοι θα είναι στην Κύπρο το Σαββατοκύριακο, εγώ θα, πάω μάλιστα το, το Σάββατο το πρωί στην Κύπρο για τη διάσκεψη των Προέδρων ε, που θα γίνει στην Κύπρο για τον εορτασμό της 20ης επαιτίου από την εσωτερική αγορά. Θα είναι αρκετά φορτωμένη εβδομάδα. Ελπίζω να την ε, εκμεταλλευτούμε και να την αξιοποιήσουμε όλοι πλήρως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάλκολ. And our Is there any other issues to be announced or any other way how we could... Uh, Τίποτε άλλο. Εν αναμονή της συγκεκριάς μας. A bit of it on, on, on the use. Συνήθως ε, δεν μας ε, φτάνει ο χρόνος, αλλά τώρα μας περισσεύει λίγο. το Αμερικανικό Επιμολυντήριο, το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δώσει μια διάλεξη για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου και που περιλαμβάνει και πολλές μελέτες και για την εσωτερική αγορά, την ενέργεια, τους σιδηροδρόμους, τα φάρμακα και τον ενιαίο χώρο ε, για τις πληρωμές. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμα αυτά τα έγγραφα και πληροφορίες. Ένα άλλο θέμα είναι οι μεταφορές μεταξύ των επιχειρήσεων, γιατί οι επιχειρήσεις που επαιδείουν στην Ευρώπη ενδιαφέρονται για εύκολες μεταθέσεις του προσωπικού τους. Σω θα πρέπει κάτι τέτοιο να το είχαμε περιλάβει στην πρόσφατη έκθεση κυρία Μπάστο, γιατί θα ανακύψει και αυτό το θέμα. Ένα άλλο ζήτημα αφορά το κέντρο για τις ευρωπαϊκές μελέτες που εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Οι, εφ... οι εφαρμογές στην ενιαία αγορά». Η εφαρμογή των διατάξεων της ενιαίας αγοράς. Και όσοι μας παρακολουθούν από το ίντερνετ μπορούν να το βρουν το βιβλίο αυτό στην ιστοσελίδα μας για την εφαρμογή των διατάξεων της ενιαίας αγοράς. Μάλιστα, κάνω και εγώ μια εισαγωγή στο, κύμα, στο έγγραφο αυτό. Και εσύ, Παύλο, φαντάζομαι θα έχεις κάποιες ιδέες. Μία ερώτηση. Θα το στείλετε στα γραφεία μας ή θα πρέπει εμείς να το ψάξουμε. Το βιβλίο της Αμερικανικής Πρεσβείας, του Αμερικανικό Επιμελητήριου και το άλλο που μας είπατε, πού θα το βρούμε. Εγώ το βράδυ θα πάω στην Αμερικανική Πρεσβεία, θα εξασφαλίσω αντίγραφα για όλα τα μέλη της Επιτροπής. Και το βιβλίο αυτό που σας ανέφερα πριν από λίγο θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΣ. Λυπούμε που βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Μόλις θα έχετε τον εξοπλισμό σας ε, έτοιμο και θα είσαστε σε θέση να ξεκινήσετε, θα ήθελα να σας δώσω τον λόγο για την τροποποίηση των επαγγελματικών όρων και προϋποθέσεων επαγγελματικών προσόντων μπορείτε να δεν πιέζει τόσο πολύ ο χρόνος ώστε να βιαστούμε τόσο και να σας ε, πιέσουμε και να μην μπορείτε να πάρετε ανάσα λοιπόν βολευτείτε πρώτα και μπορείτε μετά αφού έχετε βολευτεί να ξεκινήσετε έχετε τον λόγο Excusez-moi, συγγνώμη. Τρέχω συνέχεια σήμερα. Είναι μία από τις μέρες που με το που θα τελειώσει ίσως χρειαστεί και ακόμα. Πραγματικά είναι από τα πιο ε, λεπτά ζητήματα που χρειάστηκε να χειριστώ για την οδηγία αυτή. Ε, είχα συνάντηση με μια ομάδα νέων από την ε, περιφέρειά μου που θα, περάσουν, θα δώσουν εξετάσεις για ε, το απολυτήριο για τεχνικά επαγγέλματα και είχαν πολλές απορίες για το θέμα αυτό. Περνάω λοιπόν στο θέμα που σας ενδιαφέρει. Δεν πρόκειται να αναφερθώ σε θέματα που θίξαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση γιατί νομίζω ότι είχαμε κάνει μια αρκετά γενική και πλήρη επισκόπηση. Προτιμώ το χρόνο μας να τον αφιερώσουμε στη συζήτηση και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε για να απαντήσει στις απορίες μας γιατί στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν είχε καθόλου χρόνο ε, για ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα πάντως να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία για τα οποία θα ξανακαταθέσω τροπολογίες για μερικές διευκρινήσεις γιατί είχαμε και κάποιες εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά τη μερική πρόσβαση. Σε ό,τι αφορά τη μερική πρόσβαση, θα πρέπει να διευκρινίσουμε το γεγονός ότι αν ένα κράτος μέλος μπορεί καταρχήν να εμποδίσει την εφαρμογή της ε, μερικής πρόσβασης σε ορισμένα επαγγέλματα για ε, λόγους, ε, επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. Αυτό θα πρέπει να προεξοφλεί τη δυνατότητα των εθνικών αρχών αυτού του κράτους να παρεκκλίνω από την αρχή αυτή αν το κρίνουν σκόπιμο μετά από μια περιπτωσιολογική ανάλυση. Ε, για το θέμα αυτό φαντάζομαι θα χρειαστεί συζήτηση. Σε ό,τι αφορά την ε, εξακρίβωση των γλωσσικών προσόντων. Επαναλαμβάνω την πρόταση που έκανα την προηγούμενη φορά. Κατά τη γνώμη μου δεν ε, χρειάζεται να διευκρινίσουμε τους όρους στην άσκηση της, της επαγγελματικής δραστηριότητας και όχι ε, στη, στις γλωσσικές δεξιότητες. Γιατί το άρθρο 53 εμπίπτει στον, στο τίτλο 4 που καλύπτει τους τρόπους άσκησης του επαγγέλματος. Τώρα, αν ο έλεγχος ε, των γλωσσικών δεξιοτήτων θα πρέπει να εμπίπτει στο, στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, αυτό δεν εμποδίζει τις, ε, τους πρακτικούς τρόπους εφαρμογής και τη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών, αρκεί ο έλεγχος αυτός να είναι ανάλογος, μη συστηματικός και φυσικά να μην δημιουργεί ένα αποτρεπτικό κόστος για τον επαγγελματία, κάτι που θα δημιουργήσει έμεσο φραγμό ή και καλυμμένο εμπόδιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 35, 37, 40 και 75 που αφορούν τις συμπληρωματικές προϋποθέσεις. Οι τροπολογίες αυτές προκάλεσαν κάποιες ανησυχίες, γιατί προσθέτουν κάποιες επιπλέον απαιτήσει που ίσως φαίνονται δυσανάλογες και καταστήσουν πιο άκαμπτο το σύστημα. Και εδώ θα προτείνω κάποιες αλλαγές για να λάβω υπόψη και να διασκεδάσω τους φόβους αυτούς που τους θεωρώ και εύλογους σε τελική ανάλυση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το βασικό θέμα των οδηγιών, τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Έχουμε το πρόβλημα της μετάβασης στη δεκαετία για τις απαιτήσει σπουδών για τον πρώτο κύκλο σπουδών των νοσοκόμων. Τους τελευταίους ε, μήνες, ε, εβδομάδες μέχρι και μέρες έχω συναντηθεί με πολλούς εκπροσώπους του ενδιαφερόμενου κλάδου και κυρίως ε, εκπροσώπους το νοσηλευτικό προσωπικό από τη Γερμανία και θα ήθελα να πω ότι κατανοώ πλήρως τις ανησυχίες τους. Πάντως είχα ήδη προσπαθήσει να προτείνω μια λύση με μεταβατική περίοδο. Διαπιστώνω όμως ότι δεν αρκεί η λύση αυτή για τη μεταβατική περίοδο. Οπότε θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες και ήδη προσπαθούμε να καταλήξουμε στις συμβαστικές προτάσεις για να λάβουμε υπόψη την παράλληλη λειτουργία δύο συστημάτων με κάποιες κοινέ απαιτήσει προσόντων και δεξιοτήτων. Πάντως αυτό που διαπίστωσα μέχρι σήμερα δεν είναι επαρκείς αυτές οι προτάσεις, ούτε ικανοποιητικέ απόλυτα. Δεν είμαι εξορισμού κατά μια λύση που θα στηρίζεται στις δεξιότητες και τα προσόντα, σε ένα κατάλογο δηλαδή προσόντων. Αλλά μια τέτοια λύση είναι χρονοβόρα, γιατί αποκλείεται να προλάβουμε μέσα σε ένα ή δύο μήνες ε, να ενημερώσουμε ένα τέτοιο κατάλογο προσόντων και δεξιοτήτων, ε, ενώ ο αντίστοιχος προηγούμενος κατάλογος λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια. Και αυτό το ιατρικό επάγγελμα έχει εξελιχθεί, γιατί έχουν αλλάξει και ανάγκες των ασθενών, ε, οι τεχνολογικές ε, ανάγκες επίσης και οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν απαραίτητη την πρόβλεψη και νέων προσόντων και δεξιοτήτων για τις νοσοκόμες και το νοσηλευτικό προσωπικό. Άρα παρόν κατάλογος δεν είναι ε, ενημερωμένος. Μέσα σε 10 χρόνια ο κλάδος ε, μπορεί να υπάγεται μόνο σε ένα ε, ε, καθεστώς εξαίρεσης ειδικό και όχι σε αντίστοιχο ε, αντίστοιχη ρύθμιση, γιατί κάθε κράτος, άσχετα από το αν θα δημιουργήσουμε τελικά δύο παράλληλα συστήματα, μπορεί να εφαρμόσει διακριτική μεταχείριση και άνηση μεταχείριση μεταξύ του προσωπικού. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι κάθε χώρα μπορεί να θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνει προσπάθεια και να εναρμονιστεί σε μία εναρμόνιση προς τους πιο απαιτητικούς ρόλους και ως εκ τούτου θα καταλήξουμε σε ένα επίπεδο κατάρτισης που θα είναι λιγότερο απαιτητικό και πιο φθηνό και μάλιστα σε μια περίοδο χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης το επιχείρημα του κόστους ίσως ε, χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από τις διάφορες χώρες. Και νομίζω ότι εκεί θα απομακρυνθούμε από τη φιλοδοξία μας για εναρμόνιση προς τα πάνω. Γιατί όπως σας είπα, συζήτησα με νέους που μου, που μου είπαν ότι περιμένουν από την Ευρώπη μια ασφάλεια, μια εγγύηση και προστασία ε, μια ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μια δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, στην εσωτερική αγορά, αλλά όχι θέσεις εργασίας πάση θυσία και ε, χωρίς ποιότητα. Θα συνεχιστούν λοιπόν οι συζητήσεις. Έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο μέχρι, που, μέχρι να καταλήξουμε στη συμφωνία στις διάφορες χώρες και στα θεσμικά όργανα το Κοινοβούλιο τάσεται μάλλον υπέρ μια εναρμόνιση προς τα πάνω, προς τις πιο απαιτητικέ προποθέσει, Μετά την κατάθεση των τροπολογιών, μετά τη διορία τη 15 η Οκτωβρίου και μετά τη μετάφραση που θα γίνει των τροπολογιών, θα διοργανώσω τρεις συναντήσεις των εισηγητών και των σκιωδών βλέπω να διαμαρτύρονται οι δισκιώδεις, αλλά νομίζω ότι θα χρειαστούμε τρεις συσκέψεις μεταξύ μας πριν περάσουμε στην ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Και προειδοποιώ ήδη από τώρα τον Πρόεδρο, γιατί δεν πρόλαβα να το συζητήσω προηγουμένως μαζί του, και προειδοποιώ και τη Γραμματεία, ότι αν μετά τις τρεις συνεδριάσεις με τους σκιώδεις ηγητές, όπου φυσικά κάθε ενδιαφερόμενος ευρωβουλευτής είναι πρόσδεκτος ε, να στείλει ε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις προτάσεις ε, και τις λύσεις που προτείνει. Αλλά δεν σας εγγυώμαι ότι θα είμαστε έτοιμοι για, στη, για τις 28 Νοεμβρίου, για την ψηφοφορία δηλαδή στην ΙΜΚΟ. Για ένα όμως τόσο σημαντικό θέμα που αφορά εκατομμύρια εργαζομένων και που αφορά το αυριανό όραμα ουσιαστικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Αγορά, για την νέα εποχή, για τον 21ο αιώνα, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε ε, και λίγο παραπάνω χρόνο, έστω και αυτό σημαίνει παράταση του χρονοδιαγράμματός μας. Πάντως με ενδιαφέρει η αγαστή συνεργασία και με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Μάλιστα την επόμενη εβδομάδα το Συμβούλιο θα έχει σημαντικό, σημαντική συνεδρίαση και εκπρόσωπος ε, της Προεδρίας θα έρθει αμέσως μετά για να το συζητήσουμε είναι, επαναλαμβάνω, πολύ αρμονική συνεργασία μεταξύ των κοινωτικών θεσμικών οργάνων και ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε ικανοποιητική λύση. Thank ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στους Σκιώδη τώρα. Η κυρία Λεγκρίπ πρώτη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Βερνιό για τις διευκρινήσεις τις οποίες μας έδωσε πάνω στα τόσο σημαντικά θέματα τα οποία περιλαμβάνει η συγκεκριμένη έκθεση. Άκουσα προσεκτικά λοιπόν αυτά που μας είπατε. Ακούσατε κι εσείς αυτό το οποίο εμείς σαν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζητήσαμε να υπάρξουν περισσότερες εξηγήσει για την άρνηση μερικής πρόσβασης κατά περίπτωση. Υπάρχει εδώ μια ισορροπία ε, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί, αλλά είναι αλήθεια ότι έχουμε καταφέρει να κάνουμε σημαντικά βήματα και θα συμφωνήσουμε, είμαι βέβαια, σε κάποιες μικρές βελτιώσεις της αρχικής πρότασης την οποία μας προτείνατε και η οποία βρίσκεται στη γραμμή της έκθεσης Μακάρτιν, κάτι το οποίο θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Ευχαριστώ λοιπόν για τις διευκρινήσεις, είναι προς την καλή κατεύθυνση, στη σωστή κατεύθυνση. Άκουσα επίσης ε, αυτά που λέγατε για κάποιες από τις τροπολογίες σας Πράγματι θα πρέπει να κατανοήσουμε το σκεπτικισμό που εκπέμπουμε σαν ομάδα εμείς με τις 35, 37, 43 και 65 που εν πολλής ε, θα ε, τροποποιήσουν, όχι σε πολύ μεγάλο βάθος. Σας παρακαλώ να αντιδράσετε στις τροπολογίες αυτές ε, γρήγορα, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε από κοινού να κάνουμε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις ε, γύρω από τις τροπολογίες αυτές οι οποίες δημιουργούν ορισμένες ανησυχίες. Τώρα για το, ε, ε, για το εκλεκτό επάγγελμα των νοσοκόμων ανδρών και γυναικών. Σας ευχαριστώ για τον πραγματισμό και την κατανόηση που χαρακτηρίζουν την εργασία σας από την αρχή. Είμαι σίγουρη πως ε, με κάποια καλή βούληση από τις δύο πλευρές και με λίγο επιπλέον χρόνο θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε από κοινού τους τρόπους έτσι ώστε να συμβιβάσουμε τις διαφορετικές καταστάσεις και τα διαφορετικά συστήματα τα οποία επικρατούν σε χώρες ε, γύρω από το θέμα των νοσοκόμων και την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο σύστημα κατάρτισης. Δίνουμε μεγάλη σημασία στο αξιόπιστο σύστημα κατάρτισης και εκπαίδευσης, ένα σύστημα το οποίο για μας σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ε, είναι γενικό και ακαδημαϊκό, αλλά είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο και έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ε, έτσι ώστε να δώσουμε την δυνατότητα στην ευρωπαϊκή νεότητα να προοδεύσει. Λοιπόν, δεν θα επιμείνω. Θέλω να χαιρετήσω για μια ακόμη φορά την σημαντική προσπάθεια και του ΣΒΑΜ και άλλων συναδέλφων. Έχουμε σχεδόν καταλήξει και σχετικά με το άρθρο 31. Απαιτείται να υπάρξει μια ισορροπημένη θέση η οποία δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προβλήματα ούτε στο επάγγελμα του νοσοκόμου, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την αξιοπρέπεια και την οποία αξίζει αυτό το επάγγελμα και γι' αυτό απαιτείται και ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και προετοιμασίας και εδώ θα χρειαστεί να διατυπώσουμε με διαφορετικό τρόπο το άρθρο 31. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τελειώνοντας, με ένα επάγγελμα για το οποίο έχει υπάρξει αρκετή θα έλεγα προσοχή και έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις και προς τους εισηγητές και προς τους σκιώδεις εισηγητές και προς πολλά μέλη. Είναι το επάγγελμα του συμβολιογράφου. Η εισηγήτρια με κατάλαβε από την αρχή της φράσης μου. Στην παρούσα φάση είμαι σύμφωνη μαζί σας, κυρία Βερνιό. Νομίζω ότι και στην περίπτωση των συμβολιογράφων θα πρέπει νομίζω να καταλήξουμε στην πιο ικανοποιητική δυνατή συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λοιπόν θα προσπαθήσει να δώσει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις για την φύση των στάζ, Υπάρχει σε αυτήν την αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας η δυνατότητα αναγνώρισης των στάζ που έχουν γίνει σε άλλες χώρες και γι' αυτό θα θέλαμε να διευκρινίσουμε καλύτερα και να εμβαθύνουμε περισσότερο στην έννοια του στάζ, αναφερόμενη επίσης και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ποιότητα των στάζ που είχαν προταθεί και γίνει δεκτά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού φόρουμ για την νεότητα. Δεν θα ήθελα να σας καθυστερήσω άλλο. Με την εισηγήτρια μοιραζόμαστε πολλές απόψεις, αλλά υπάρχουν κάποιες προσπάθειες που πρέπει να γίνουν ακόμα από κοινού. Η κυρία Ρίλε των Πρασίνων, ναι, ευχαριστώ. Δυστυχώς, δυστυχώς δεν παρακολούθησα την παρέμβαση της εισηγήτριας, ζητώ συγγνώμη. Έχουμε πολλά θέματα που παρακολουθούμε πέρα από τα προσόντα για τα επαγγελματικά προσόντα έχουμε και τα άλλα θέματα. Επιστρέφω στο θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Μπορώ να σας πω Οπωσδήποτε αυτά τα οποία θα κατατεθούν από δική μας πλευρά. Το είχα πει και σε μια από τις τελευταίες συζητήσεις ότι τον τομέα της μη ακαδημαϊκής, μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλαδή τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάτησης θέλουμε να τον προωθήσουμε από την αμυντική θέση να περάσουμε σε πιο επιθετική θέση τη σημασία της διπλής, διτής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αναφέρεται πολλές φορές αλλά δεν, έχει, δεν βρίσκει αντανάκλαση και ισοδύναμο στις νομικέ προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι θα υποβάλουμε εμείς κάποιες προτάσεις σχετικά. Επίσης θα αποσαφηνίσουμε για άλλη μια φορά ότι το επαγγελματικό πιστοποιητικό πρέπει να είναι εθελοντικό, εθελούσιου χαρακτήρα. Έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να πιέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να επιβάλλει ένα άλλο πρότυπο Πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευόμαστε τις συλλογικές, ε, τις ενώσεις συλλόγους επαγγελματιών προτού προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι αυτονόητο ότι η χώρα <clears throat> προέλευσης δεν μπορεί να αναγνωρίζει αυτά τα θέματα, αλλά μπορεί να υποβάλει και να προετοιμάζει αυτά τα θέματα και να τα πιστοποιεί η χώρα προέλευσης, αλλά η αναγνώριση πρέπει να γίνεται από τη χώρα υποδοχής, εκεί όπου θα παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Και αυτό δεν το αποσαφηνίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν κάποια σύγχυση εδώ, συγχέονται κάποια πράγματα. Και όσον αφορά και την πρόσβαση ε, σε σχέση με τους ασθενείς, πάει, ε, ακολουθεί διαφορετική πορεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει ότι το κράτος προέλευσης μέρος, τμήμα ενός ε, τέτοιου επαγγέλματος μπορεί να το καλύπτει ή να το αναγνωρίζει και στην άλλη χώρα θα πρέπει ε, να μπορεί να ίσως να μην αναγνωρίζεται κάτι τέτοιο ή να υπάρχει κατακαιρματισμός. Αυτός ο κατακαιρματισμός όμως ε, των επαγγελματικών αυτών προφίλ, των εικόνων αυτών επαγγελμάτων δεν είναι κάτι θετικό και βρίσκω ότι είναι προβληματικό αν τέτοιου είδους επαγγέλματα εκ των έξω προσπαθεί κανείς να τα κατακαιρματίσει. Δεν ήταν αυτό το θέμα της πρόσβασης για την περίθαψη των ασθενών ε, από νοσοκόμους και προσπάθησα να το αποσαφηνίσω. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα γραφειοκρατικής επιβάρυνσης, γραφειοκρατικό επαχθές βάρος προκαλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει εδώ και σε σχέση με τον ενιαίο ομόλογο ή εταίρο, διαρωτώ με γιατί δημιουργούνται προβλήματα. Όλα αυτά οδηγούν σε υπερβολικές ε, γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, με διαφορετικές αρμοδιότητες από πλευράς διαφορετικών αρμόδιων. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα που είναι σκόπιμα και αναγκαία. Και αν έχουμε έναν ενιαίο ομόλογο εταίρο, τότε τίθεται το ερώτημα γιατί πρέπει να δημιουργηθούν περαιτέρω θηρίδες ή και άλλοι αρμόδιοι στο θέμα της ε, χρονικής περίοδου, time period, για τις χρονικές προθεσμίες, θα πρέπει να τα ξαναδούμε τα πράγματα. Τα είδαμε εμείς και είμαστε κατά της ε, ε, ε, ε αναγνώρισης Πιστεύουμε ότι αυτά τα σημεία ναι μεν πρέπει να μπορέσουν να καλυφθούν, αλλά πρέπει να αποσαφινιστεί ότι μόνο επιπρόσθετα μπορούν να αναφέρονται, δεν μπορούν να είναι υποκατάστατα όσον αφορά ε, προδιαγραφές και διατάξεις ε, ε, γιατί θα πρέπει να δούμε δεν υπάρχει ένας εναρμονισμένος ορισμός μέσω της διαδικασίας Μπολόνια απέρευσαν πολλά πράγματα και δεν είναι με βάση μια ενιαία νομοθετική ρύθμιση μόνο επιπρόσθετα μπορούν να λειτουργήσουν και όχι ως υποκατάστατα και έχουμε καταθέσει και τροπολογίε για αυτό το θέμα. Έρχομαι στο τελευταίο σημείο. Προσπαθώ να είμαι σύντομη όσο γίνεται. Έχουμε φυσικά προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε όσον αφορά τι αδελφέ νοσοκόμε. Σίγουρα πιστεύω ότι πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε εδώ να καθορίσουμε σαφώς τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες όμως ε, δεν μπορεί να καθοριστούν αυτά μόνο με τον αριθμό των ετών σχολικής εκπαίδευσης. Γι' αυτό έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες και πιστεύω ότι με τους φαρμακοποιούς ε, το παλαιό καθεστώς πρέπει να αποκατασταθεί. Δεν κατανοώ τη διαγραφή, την απάλληψη που έγινε. Τελευταίο σημείο για τις τροπολογίες. Κάπως δυσάρεστη εντύπωση έχω, όχι μόνο διότι έχει πολλές κατεξιοδότηση πράξη η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπει, αλλά και τη διαβούλευση την έχει έχει περιορίσει. Τα παλαιά άρθρα τα έχει διαγράψει εντελώς και αντικαθίσταται από ένα νέο άρθρο το οποίο αποκαλείται λέει διαφάνεια. Διαφάνεια. Η διαβούλευση όμως είναι κάτι διαφορετικό από τη διαφάνεια, έτσι δεν είναι. Και πιστεύω ότι σε ένα τόσο σημαντικό πεδίο χρειαζόμαστε τη διαβούλευση και στην ομοθεσία πρέπει να αντανακλάται αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. <clears throat> And, uh... Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη μου, λίγο αφηρημένη πριν κύριε Μπουσόη. Κανονικά σε εσά έπρεπε να δώσω πρώτα το λόγο. Όχι, κανένα πρόβλημα κυρία Πρόεδρε. Ήδη είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τις θέσεις μου ε, επί της σημαντικής έκθεσης κυρίας Βερνιό για τα επαγγελματικά προσόντα, οπότε σήμερα μπορώ να περιοριστώ σε κάποια νέα θέματα. Πρώτα απ' όλα όμως να επαναλάβω την αρχική μου εκτίμηση ότι είναι καταπληκτική η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Βερνιό και θα αποτελέσει εξαιρετική βάση για τη σύναψη συμβαστικών ε, προτάσεων. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, για την ε, προσπάθεια της εισηγήτριας να γίνει πιο ελαστική στις τροπολογίες 35-37 γιατί ο περιορισμός ε, ε, στην πλήρη ε, άσκηση του επαγγέλματο του 37 ή της υποχρέωσης που προβλέπει η τροπολογία 37 που θα δυσκολεύσει κυρίως τους ξεναγούς και έτσι θα δημιουργηθούν κάποιοι φραγμοί για την ε, κινητικότητα και την ε, αναγνώριση των προσόντων. Χαίρομαι λοιπόν για την ελαστικότητα στις τροπολογίες αυτές. Ό,τι αφορά την τροπολογία 75, καθιστά την ε, αυτόματη αναγνώριση ακόμη πιο δύσκολη εφόσον δεν έχει ασκηθεί το επάγγελμα κατά μία τετραετία. Αν οι επαγγελματίε πρέπει να αποδείξουν την άσκηση αυτή, η όλη διαδικασία αναγνώριση θα γίνει πολύ πιο επαχθή. και αυτό ακριβώ προσπαθούμε να αποφύγουμε με την έκθεσή μας. Βέβαια, ξέρω ότι καταθέσατε την τροπολογία 75 για να εξασφαλίσετε την προστασία των ασθενών. Κατά τη γνώμη μου όμως, το μήνυμα που στέλνουμε την τροπολογία αυτή είναι σφαλμένο. Ας το ξανασκεφτούμε και ας προσπαθήσουμε να βρούμε άλλους τρόπους να εξασφαλίσουμε όλα τα εχέγγυα της ε, προστασίας των ασθενών. Σε ό,τι αφορά τις ε, επαγγελματικές κάρτες, θα καταθέσω τροπολογίες για να διευκρινίσω κάποιες πρακτικές πτυχές. Το θέμα είναι ποιος θα λαμβάνει την απόφαση για την θέσπιση μιας επαγγελματικής κάρτας για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Και σε περίπτωση σιωπηρής αναγνώρισης. Αυτό σημαίνει ότι ο επαγγελματίας θα έχει πρόσβαση στο επάγγελμα. Σε ό,τι αφορά τους γλωσσικούς ελέγχους και εκεί θα πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις και να δούμε πότε θα γίνονται αυτές οι εξακριβώσεις. Ίσως αυτοί οι έλεγχοι έχουν νόημα πριν να επιτραπεί η πρόσβαση του επαγγελματία στο επάγγελμα. Γιατί προ το παρόν δεν είναι σαφέ ούτε από την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε από τι τροπολογίε πότε γίνονται αυτοί ε, οι έλεγχοι, η εξακρίβωση των γλωσσικών ε, προσόντων. Επίσης, ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τις ε, νοσοκόμες ε, με βάση ε, το καθεστώς των κεκτημένων δικαιωμάτων. Είναι κάπως ιδιάζουσα η κατάσταση των νοσοκόμων από την Πολωνία και τη Ρουμανία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι νοσοκόμες αυτές που έχουν πτυχίο ή έχουν ξεκινήσει την κατάρτισή τους πριν την ένταξη των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πληρούν ε, ειδικέ προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν τα προσόντα τους. Θα πρέπει να χορηγήσουν ένα πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει ότι είχαν, την επαγγελματική, είχαν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ε, ε, πενταετή, 7 χρόνια πριν την υποβολή του αιτήματο. Άρθρο 33 και 33α τη οδηγία. Βέβαια, μετά την ένταξη, η κατάσταση στην Πολωνία έχει εξελιχθεί και προβλέπεται συμπληρωματική κατάρτιση των νοσοκόμων αυτών για να ευθυγραμμιστούμε τι απαιτήσει τη οδηγία. Οπότε δεν υπάρχει λόγος για τα περαιτέρω κριτήρια του άρθρου 33. Αλλαγές έγινε και στη Ρουμανία, γιατί η κατάρτιση των νοσοκόμων πριν το 2007 ήταν περιορισμένη ως μεταξύ. Οι νοσοκόμες αυτές έχουν συνεχίσει συμπληρωματικές καταρτήσεις και σε πανεπιστήμια ή έχουν ε, παρακολουθήσει ε, σεμινάρια για την αναβάθμιση των προσόντων τους. Άλλωστε δεν υπήρξαν περιπτώσεις ε, κατάχρησης ή κακής πρακτικής αυτών των νοσοκόμων, οπότε δεν υπάρχει ε, κανένας κίνδυνος για τους ασθενείς, ούτε χαμηλότερη ποιότητα ε, των επαγγελματικών προσόντων αυτών των νοσοκόμων. Ελπίζω και το Συμβούλιο να επαναθεωρήσει τη θέση του και να σκεφτεί κατά, κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξει η πενταετία ε, για την τελευταία, στην τελευταία επταετία να γίνει τριετία στην τελευταία πενταετία. Νομίζω ότι μια τέτοια αλλαγή για την Ρωμανία και την Πολωνία ευθυγραμμίζεται με την αρχή τη ίση μεταχείριση που αποτελεί θεμέλιο λίθο τη εσωτερική αγορά. Αυτά. Ευχαριστώ θερμά κυρία Βερνιό και ευελπιστώ ότι θα έχουμε και πολύ καλέ συμβαστικέ τροπολογίε στο τέλο. Ευχαριστώ η ΕΜΑ από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γενικά είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τις κατευθύνσεις της εισηγήτριας. Συνεργαστήκαμε νομίζω πολύ καλά. Κατέθεσα ορισμένε προτάσεις τροπολογίας που νομίζω ότι ενίσχυσαν την έκθεση και καθόρισαν καλύτερα τις τροπολογίες γύρω από το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης. Οι τοπολογίε μου έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη και την αύξηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών για τους επαγγελματίες, πάντα με συγκεκριμένες εγγύησεις. Η πιο σημαντική πλευρά αφορά τον μηχανισμό διαφάνειας. Εδώ έχω καταθέσει πολλές τροπολογίες για την τόνωση του άρθρου 59 για να μπορούμε να αναλύσουμε καλύτερα την κατάσταση των ρυθμιζόμενων τομέων στα διάφορα κράτη-μέλη να δούμε που ε, κάποιες χώρες παρεμποδίζουν ε, δυσανάλογα την ε, είσοδο σε ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες και σε ποιο βαθμό αυτό μειώνει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες ενίας αγοράς. Σχετικά τώρα με το μηχανισμό πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά, θα καταθέσω τροπολογίες για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε όταν οι επαγγελματίες έχουν περιοριστεί τα δικαιώματά τους να μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση ευκολότερα. Και φυσικά οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προτείνονται για την ασφάλεια των ασθενών στον συγκεκριμένο τομέα είναι αυστηρότατες και πολύ σωστά. Υποστηρίζω λοιπόν Νομίζω ότι θα πρέπει όμως να καλύψουμε και τους ε, εργαζόμενους στον κοινωνικό τομέα αν δεν το ρυθμίσουμε αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπλέον κινδύνους στους ασθενείς. Θα πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε βέβαιοι ότι δεν κάνουμε εισοδισμό θα έλεγα στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και σχετικά τώρα με την ανάγκη για μια επαγγελματική ταυτότητα. Αυτό έχει σημασία μόνο αν υπάρχει ένα μητρό ευρωπαϊκό πίσω ε, εγώ έχω υποστηρίξει την απόκτηση αυτής της κάρτας, αλλά σε εθελοντική βάση. θα πρέπει να γίνεται μετά από αίτημα των ιδίων των επαγγελματιών εφόσον το επιθυμούν. Η κάρτα αυτή θεωρητικά θα πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες της γραφειοκρατικές και αν δεν καταφέρνει να μειώνει όλες αυτές τις χρονοβόρες διαδικασίες θα έχει αποτύχει το σύστημα της κάρτας. Κάποιες από τις προθεσμίες τις οποίες έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ αισιόδοξε, αλλά ελπίζω να καταφέρουμε να τις αλλάξουμε. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε επίσης και τους εργοδότες να κάνουν ελέγχους όταν θεωρούν ότι είναι χρήσιμο και στην φάση της πρόσληψης των υπαλλήλων τους και κατά τη διάρκεια της άσκησης των, ε, των δραστηριοτήτων τους. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς και τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε σε σχέση με το δωρεάν καθεστώς ε, των ε, τεστ γλωσσών Και τέλος, για την μερική πρόσβαση, το πρώτο θέμα το οποίο τέθηκε από την κυρία Βέρνιο σήμερα, όταν εγώ υπέβαλα την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τη διαβούλευση, είχα μεταφέρει τις επιθυμίες γενικά πολλών επαγγελματιών και φαίνεται ότι δεν υπάρχει συμφωνία γύρω από το θέμα της μερικής πρόσβασης. Κανένας δεν έχει πει ξεκάθαρα ότι είναι υπέρ αυτού του συστήματος και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσο προσφέρει λύσεις. Ακόμα και αν υπάρχει εξαίρεση ή απόκληση αδειοδοτημένη από, για ένα κράτος μέλος, είναι ε, καλύτερα να θεωρηθεί αυτό ένα νομικό θα έλεγα προηγούμενο και κατά περίπτωση να αντιμετωπίζεται η χορήγηση της εξαίρεσης και να μην υπάρξει μια ειδική ρύθμιση ξεχωριστή ε, νομική για το θέμα της μερικής πρόσβασης. Λοιπόν, ε, έθεσα τις προτεραιότητες μου, ελπίζω να της λάβει υπόψη η κυρία Βερνιό και οι υπόλοιποι σκιώδεις. Ελπίζω να καταλήξουμε σε περαιτέρω συμβιβαστικές. Είναι απαραίτητο να βρούμε λύσεις συμβιβαστικές για τους επαγγελματίες σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει κάποιος σκιώδης. Θα δώσω το λόγο Βαντερκάμ, Σβάμπ και μετά εγώ ίδια. Ο Βαντεν Κάμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συνεχίζοντας ακριβώς σε αυτά που η αξιότιμος συνάδελφος ε, κυρία Λεγκρίπ ανέφερε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της εισηγήτριας στους όρους ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης αυτών των επαγγελμάτων των αδερφών. Τίθεται το ερώτημα στην Γερμανία και στην Ολλανδία αν θα είναι 5 ή 10 χρόνια. Προτιμώνται τα 10 χρόνια γιατί αν θα ήταν 12 πώς θα μετρηθούν, πώς θα προσμετρηθούν. Πιο απλά και πιο συνοπτικά δεν μπορώ να διατυπώσω το ερώτημα. Αν έχετε μία απάντηση επιλύεται αυτόματα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Εσείς παρακαλώ έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Μπάρβαρα Βάιλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και στην τελευταία συνεδρίαση για άλλη μια φορά θέλω να υποστηρίξω την εισηγήτρια μας στην θεμελιώδη κατεύθυνση που ακολουθεί και στους, στα, στα επιμέρους τμήματα της έκθεσής της. Έχω δύο μικρές ε, τροποποιήσεις που θα ήθελα να ληφθούν υπόψη Ίσως όμως ε, δεν μπορούν να διατυπωθούν θετικά με τις τροπολογίες. Το 34 για παράδειγμα για την πλήρη απασχόληση να αποσυρθεί και να φεθεί το αρχικό κείμενο της Επιτροπής θα ήταν ίσως το απλούστερο. Και έτσι διαπίστωσα και σε σχέση με την τροπολογία 59 επίσης ότι οι 5.000 επιθυμούμενες ώρες για τις μαμές, τις ΜΕΕΣ, δεν είναι ρεαλιστική προϋπόθεση και ίσως απλούστερο θα ήταν να επιστρέφαμε στο αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου δεν επιβάλλεται κάποιο τέτοιο όριο ορών. Θα έπρεπε να, να εξετάσουμε το αίτημα του κυρίου Μπουσόη για τις ξεχωριστές ε, απαιτήσει για τους Ρουμάνους ε, εργαζόμενους ε, που θα έπρεπε ίσως σταδιακά να προσαρμοστεί το πλαίσιο αυτό για αυτούς με το πλαίσιο που ισχύει για τους άλλους. Είμαι με ανοιχτό πνεύμα αντιμετωπίζω αυτό το θέμα, πώς θα πρέπει να επιληθεί. Θα ήθελα να ακούσω την τεκμηρίωση για αυτή την μερική πρόσβαση, όπως προαναφέρθηκε. Ουσιαστικά υπάρχει σαφή συνένεση στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό να απαλληφθεί, να διαγραφεί πλήρω. Αν πιστεύετε εσεί για νομικού λόγου ότι θα πρέπει να παραμείνει αυτό, ίσω θα μπορούσατε να το αιτιολογήσετε, να επιχειρηματολογήσετε σχετικά. Μόνο μία τροπολογία ε, Έχω αρκετές τροπολογίες, αλλά προς μία κατεύθυνση, κάπως την κατεύθυνση της κυρίας Ρούλε θέλω να κινηθώ με αυτήν. Θα ήθελα όλα αυτά που εμείς κατά την τελευταία αναθεώρηση της οδηγίας κάναμε και στην προτελευταία ακόμα σε σχέση με το διπλό, το διτό σύστημα για τους Γερμανούς χειρόνακτες για παράδειγμα, μαθητευόμενους σε χειρονακτικά επαγγέλματα. Στην τάση τουλάχιστον θέλω να καταλήξουμε σε εκείνο το επίπεδο και σε εκείνο το επίπεδο ισοδυνάμων που ίσχυε παλαιότερα. Δεν θέλω να συρρυκνωθεί αυτό ή να υποβαθμιστεί, αυτό θα ήταν μια υποβάθμιση, μια οπισθοχώρηση στη συζήτηση που δεν θα ε, μπορούσε να δικαιολογηθεί. Χαιρόμαστε για το ότι με το διπλό διτό αυτό σύστημα μπορούμε πολλούς νέους να εντάξουμε και που δεν είναι εύκολο για αυτούς να καταφέρουν να σπουδάσουν και καταλήγουν σε αυτή τη δυνατότητα. Θέλουμε αυτή η ισοτιμία, αυτή η ισοδυναμία να επιτρέπεται για αυτά τα οποία κάνουν. Τέλος, αυτό που θέλω να υποστηρίξω την τάση, κυρία Βερνιό, για τα επαγγέλματα υγείας 12 χρόνια γενικής εκπαίδευσης να προβλέπονται. Θέλω να υποστηρίξω αυτή την πρόταση. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είδα την τροπολογία της κυρίας Βάις Γκέρμπερ. Καλό θα ήταν αν θα την είχαμε την τροπολογία. Η συζήτηση στην Γερμανία θα μπορούσε κάπως πιο ευλίγιστα, ευέλικτα να διαμορφωθεί να διαμορφωθεί με λιγότερες αγκυλώσεις ας το πω έτσι ε, όπως παρουσιάζονται αυτά τα θέματα στον τύπο είναι δίσκαμπτα θα ήταν όμως μια λαθασμένη προσέγγιση αν επιχειρηματολογούσαμε στη Γερμανία και λέγαμε υπάρχουν πολύ λίγοι άνδρες και γυναίκες νέοι νέες γυναίκες και νέοι άνδρες στα επαγγέλματα υγείας και γι' αυτό δεν θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις απαιτήσει. Το αντίθετο ισχύει. Έλλειψη προσοντούχων ε, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο και μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο καθιστώντας πιο θελκτικό το επάγγελμα, χρησιμοποιώντας όλους τους πόρους για να γίνει αυτό. Ξέρουμε ότι στην Ευρώπη πάνω από ένα τρίτο αποχωρούν από το επάγγελμα οι νέοι, επειδή με το επάγγελμα το οποίο έχουν επιλέξει δεν ικανοποιούνται ούτε με τους όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης, ούτε και με την εικόνα αυτού του επαγγέλματος. Με δύο χρόνια δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα, αλλά τα δύο χρόνια αυτά θα ήταν μια καλή ευκαιρία στη Γερμανία να ξαναπροβληματιστούμε, να δούμε πώς θα αλλάξουμε το σύστημα, πώς θα το μεταβάλουμε και θα το βελτιώσουμε προς την κατεύθυνση που ακολούθησαν και οι Αυστριακοί. Αυτό θα ήταν μια καλή κίνηση για Γερμανία. Καλό θα ήταν αν παραμέναμε σε αυτό το πλαίσιο, με αυτή την προσπάθεια και μπορούσαμε να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε για αυτές τις δύο χώρες στην Ευρώπη που δεν έχουν φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Βερνιό για την ε, πολύ αξιόλογη της έκθεση, παρόλο που έχει μερικές αδυναμίες που θα προσπαθήσω να συμβάλλω και εγώ στη βελτίωσή τους. Και ο στόχος, ο θεμελιώδης στόχος που είμαστε ενωμένοι ενώπιον του είναι ότι χρειαζόμαστε μια πιο ανοιχτή ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Διότι στην δική μου περιφέρεια, όπως και το 2005 με την Επιτροπή Ενίας Εσωτερικής Αγοράς, όπως τα είδαμε, στην δική μου εκλογική περιφέρεια μέχρι το 2020 λείπουν 500.000 θέσεις απασχόλησης ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις σημερινές έστω ανάγκες που υπάρχουν. Δηλαδή βρισκόμαστε μπροστά σε ε, υπαρξιακές ανάγκες επιβίωσης, ε, ανάγκες πραγματικής επιβίωσης και όπως αναφέρει και ο Επίτροπος 85% των Ευρωπαίων είναι ικανοποιημένοι στην περιφέρεια στην οποία ζουν παρότι δεν βρίσκουν δουλειά εκεί έστω. Με αυτή την οδηγία όμως πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα ώστε η πολυμορφία της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη να είναι το, πιο το δυνατόν πιο ανοιχτή και να επιτυγχάνεται όσμωση. Δεν είναι εύκολο αυτό. Έχουμε διαφορετικές παραδόσεις, κανόνες ε, στα κράτη-μέλη και δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τους συναδέλφους από άλλες χώρες, αλλά διαφωνώ μαζί σας κυρία Βάιλερ. Δεν θέλουμε να ικανοποιήσουμε κανένα ξεχωριστά. Θέλουμε μια ανοιχτή αγορά εργασίας. Αναζητούμε ειλικρινά και ανοιχτά συμβιβασμούς. Και για την διπλή, διτή εκπαίδευση και κατάρτιση, όπου μαθαίνει κανείς σε μια επιχείρηση αυτά τα οποία χρειάζεται, αυτές τις δύο δυνατότητες ε, για εκπαίδευση πρέπει να τις έχουμε παράλληλα. Και δεν είναι κάτι που ισχύει μόνο στην Αυστρία Γαλλία, Γερμανία ή Ολλανδία. Παντού στην Ευρώπη θα έπρεπε να είναι αυτό εφικτό και δυνατό. Παντού υπάρχουν νέοι που χρειάζονται συγκεκριμένε κατευθύνσει, χειρονακτικέ ή μια μαθητείας για να μπορέσουν να κερδίζουν χρήματα από ένα επάγγελμα στο οποίο θα καταλήξουν. Δεν πρέπει να είμαστε περιοριστικοί. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να αφήσουμε ανοιχτή αυτή τη δυνατότητα για όλου αν γίνεται. Θα χαιρόμουν αν, όπω το είπε η κυρία Λεγκρίπ, είχαμε μια νέα αναδιατύπωση του άρθρου 31, όπω. από κοινού την εξεπώνησα με την συνάδελφο Βάις Γκέρμπερ. Δεν είναι όλα τέλεια. Στο τέλο όμω μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Δεύτερον, η μερική πρόσβαση σε επαγγέλματα. Είναι σαφέ ότι υπάρχουν επαγγέλματα που υπό το πρίσμα τη Επιτροπή καθιστούν αναγκαία μια γενική ρύθμιση για αυτά. Εσεί το αναφέρατε, Πρόεδρε, ότι τα κράτη-μέλη σε επιμέρου περιπτώσει μπορούν να απορρίπτουν αυτή την μερική πρόσβαση και πάντα με βάση του τι ισχύει για την εκπαίδευση αυτή ή το επάγγελμα αυτό στην χώρα προέλευσης. Εγώ όμως θα επιθυμούσα σε ένα αιτιολογικό, να πούμε σε μια αιτιολογική σκέψη να πούμε ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη εφόσον μπορεί να επιτευχθεί αυτό από αυτή την μερική ε, πρόσβαση να κάνουν χρήση ως δυνατότητα. Να μην πούμε στο άρθρο αυτό ότι μπορούν να απορρίψουν τα κράτη-μέλη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά να λέμε ότι σε επιμέρους περιπτώσεις μπορούν να επιτρέπουν τα κράτη-μέλη κάτι τέτοιο, ώστε να αφήσουμε ένα ε, περιθώριο ελιγμών για τα κράτη. Τρίτον, οι συμβολεογράφοι από αυτό το πεδίο πλήρως εξαιρούνται σε σχέση με αυτήν την οδηγία. Σε εμά όμω από τον συνάδελφο Καράς και εγώ συμμερίζομαι την άποψή του υπάρχει επιθυμία που, για τους συμβολεογράφους που καλυπτόντουσαν μόνο από το πρωτογενές δίκαιο να τους καλύψουμε και αυτούς εδώ σε αυτό το πλαίσιο και να του δώσουμε την αναγκαία προστασία που χρειάζονται. Αλλά μην του εξαιρέσουμε απόλυτα από την εσωτερική αγορά σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών που, έχουν, που προβλέπεται υποχρεωτική έδρα ανοίγοντας τη δυνατότητα για τους ε, ε, συμβολεογράφους να έχουν μια ενδιάμεση θέση μεταξύ της δικής σας πρότασης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξευρεθεί ένα συμβιβασμός. Υπάρχει ένα άλλο σημείο το οποίο δεν αναφέρθηκε που σύντομα θα ήθελα να το αναφέρω. Αφορά το θέμα πώς καταλήγουμε σε επαγγελματικά τέτοια πιστοποιητικά. Αναφέρθηκαν κάποια πράγματα από την κυρία Ρούλα. Αν υπάρχουν τέτοια πράγματα θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα πανευρωπαϊκά, διαφορετικά δεν τα χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι το σημαντικό ερώτημα για μένα ποιο είναι εκείνο που μπορεί να δημιουργεί ένα τέτοιο επαγγελματικό δίπλωμα αναγνώριση. Είναι οι επαγγελματικέ ενώσει και σύλλογοι. Αν ναι, ποιε και πόσε και ποιοι και πόσοι, από ποια κράτη-μέλη. Να γνωρίζουμε σαφώ ποιο στο τέλο μπορεί να ζητήσει να εκδοθεί και να υπάρχει ένα τέτοιο επαγγελματικό επαγγελματικό πιστοποιητικό. Αναφέρθηκαν αρκετά για του φαρμακοποιού. Νομίζω ότι με καλή συνεργασία στο τέλο θα καταλήξουμε σε θετικέ λύσει. Ευχαριστώ για την προσοχή. Thank you. Then on my behalf I would like to, uh, Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή της δουλειά. να της πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσει όχι μόνο διαφορετικές σκέψεις, όχι μόνο διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις, αλλά και πάρα πολλές εθνικές πρακτικές οι οποίες είναι μεταξύ τους ε, δύσκολα συμβατές. Θα ήθελα να θέσω και εγώ κάποια από τα θέματα τα οποία προσωπικά θεωρώ πολύ ευαίσθητα και σημαντικά. Πρώτον, σε ορισμένες περιπτώσεις έχω επιφυλάξεις για την αυτόματη αναγνώριση για διάφορα ευαίσθητα επαγγέλματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ελπίζω να μπορέσουμε να δούμε πάλι και κάποιους από τους ορισμούς να τους αναπτύξουμε καλύτερα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται να είμαι τόσο υπέρ της ε, ελεύθερης αγοράς. Πρόβλημα έχω επίσης και με την επιμέρους πρόσβαση σε ένα επάγγελμα, τη μερική πρόσβαση. Ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε ήδη πάρα πολύ αφορά ε, τα επαγγελματικά προσόντα των νοσοκόμων. Εγώ είμαι υπέρ της 12 ετίας. Είναι προς το δικό μας εθνικό συμφέρον θα έλεγα. Υπάρχουν όμως και διαφορετικές προτάσεις, ελπίζω όμως να σας πείσουμε. Το θέμα το γλωσσικό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και τη χρήση της, των πλέον διαδεδομένων ευρωπαϊκών χωρών πολλές φορές φαίνεται ότι έχει μεγάλη σημασία το θέμα το γλωσσικό. Ευχαριστώ πάντως για την προσπάθεια την οποία έκανες και για τις προσπάθειες για να βρεθούν συμβιβαστικές λύσεις. Θα ήθελα τώρα να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Είναι η δεύτερη φορά που τίθεται υποσυζήτηση αυτό το χαρτοφυλάκιο. Καλωσορίζουμε θερμά την έκθεση κυρία Βερνιό. Ιδιαίτερα το σημείο για το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο, Επαγγελματικό Διαβατήριο, Professional Card. Είναι μια ιδέα από αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή που έδωσε συνέχεια σε αυτήν ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Και είναι καλό να υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο συνάφειας της πολιτικής εδώ, στο τέλος να μπορέσουμε να πετύχουμε μια απλούστευση με το μέσο στο οποίο θα καταλήξουμε. Αν είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα στο τέλος, με μεγαλύτερες περιόδους, εδώ άλλο πρόβλημα, αλλού άλλο, ε, τότε δεν θα καταφέρουμε να πάμε μπροστά. Δεν θα καταφέρουμε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες αναγνώρισης προσόντων. Για μας ε, το θέμα της ε, ε, εντολής αδειοδότησης είναι σημαντική απλούστευση. Να είμαι πιο σαφής. Πρώτον, η σιωπηρή αυτή αναγνώριση, η σιωπηρή αυτή αποδοχή δεν ε, είναι κάτι το οποίο απλά σημαίνει ότι κάποιος ε, μπορεί να αρχίσει να δουλεύει. Είναι μια σιωπηρή αναγνώριση διπλώματος και με τις ε, εξετάσεις τις γλωσσικές που πρέπει να γίνουν ένα θέμα θέλω να αναφέρω και θέλω να το υπενθυμίσω. Τα επαγγελματικά προσόντα είναι κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με το Solvit System 40% των περιπτώσεων Solvit συνδέονται με ένα πρόβλημα. Το ότι οι αρμόδιες αρχές δεν αντιδρούν και δεν κάνουν εκείνο το οποίο πρέπει στο τέλος θα σας πούν ότι δεν μας δίνεται απάντηση μέχρι τέσσερις μήνες. Παίρνει έξι μήνες ε, κάθε χρόνο ή και παραπάνω για να δοθεί απάντηση. Υπάρχει ε, κατεπίγουσα ανάγκη να υπάρξει ένας μηχανισμός που θα εξευρεθεί ώστε τα κράτη-μέλη να αναγκάζονται, να οδηγούνται στο να απαντούν νωρίτερα. Αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Πρέπει να συνεισφέρουμε να αποσαφινιστεί αυτή η αρχή και να λειτουργήσουν τα πράγματα σε διαφάνεια ώστε να αποφευθεί νομική αβεβαιότητα, να μην νομίζει ο ένας γιατρό ότι μπορεί άμεσα ή τέλο πάντων κάποια χρονική στιγμή να αρχίσει να εργάζεται χωρίς όλα να έχουν προετοιμαστεί. Προσπαθώ λοιπόν να είμαι σύντομο. Ε, προσωρινή κινητικότητα, temporary mobility και αναφέρομαι στι τροπολογίε 35, 37, τροπολογίε 40 και ε, συναφήσει και ερωτήματα σε σχέση με την κυρία Λεγκρίπ σε προηγούμενη συζήτηση. Οι κανονισμοί διατάξεις ε, για την κινητικότητα είναι σχετικά καινούργιοι όσον αφορά την οδηγία αυτή. Τώρα, αν θέλει το Κοινοβούλιο να αλλάξει αυτές τις διατάξεις, αυτή η αλλαγή θα γίνει σε πολύ μικρή πιεστική χρονική περίοδο, σε ένα-δύο χρόνια. Γι' αυτό είμαστε πολύ πιο συνετοί, πολύ πιο επιφυλακτικοί σε σχέση με αυτό το θέμα. Για αυτές τις τρεις τροπολογίες είχαμε θέματα και άλλα επίσης. Η περίπτωση ενός εκπαιδευτή ε, σκι ε, χιονοδρόμου που δεν θα μπορούσε να δώσει μαθήματα ε, σε μια χώρα ή στην Ιταλία ή αλλού και πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Το ίδιο αναφέρεται και με πλήρους απασχόλησης εργαζόμενους ή με εποχικής εργασίας εργαζόμενους. Να σκεφτεί κανείς ε, πόσοι μετακινούνται μεταξύ ε, Παρισίων και Βρυξελών ε, ή Βρυξελών και Κολονίας. Τι θα γίνει, θα εξαιρούνται αυτοί από την προσωρινή κινητικότητα. Επίσης, τροπολογία 40 για την ασφάλιση. Ήδη υπάρχει υποχρέωση να αντανακλάτε το θέμα της ασφάλισης στην οδηγία. Γιατί να πάμε πιο πέρα από αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει συνεισφορά για τη μελλοντική συζήτηση όταν θα υπάρχουν οι τροπολογίες. Μερική πρόσβαση. Μερική πρόσβαση ερώτημα της κυρίας Βάιλερ. Ο κυριότερος λόγος αυτό δεν είναι κάτι που επινοήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε νομολογία του 10 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και όλο και περισσότερες περιπτώσεις συσσωρεύονται. Έχουμε και προσφυγές για ε, τα επαγγέλματα υγείας και το ερώτημα επίσης ποια επαγγέλματα είναι αυτά τα οποία εμπλέκονται εδώ για την κινητικότητα, αλλά και οι μηχανικοί και οι μηχανολόγοι ιδιαίτερα ενδιαφέρονται σε σχέση με αυτά τα θέματα. Αυτό θα πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Αν δεν υπάρχει σαφήνεια από πλευρά κειμένου, με χαρά να δούμε τροπολογίες που θα συνεισφέρουν να αποκατασταθεί η διαφάνεια. Τώρα εκπλήσωμε κάπως γιατί οι μηχανολόγοι ε, είναι ε, τόσες πολλές οι προσφυγές αυτών και όχι π.χ. των αρχιτεκτώνων. Ίσως μπορούν αυτά όλα να διευθετηθούν. Χρειάζεται απολύτως νομική βεβαιότητα σε σχέση με τέτοια θέματα έναντι π.χ. Ε, θεμάτων που μπορεί να καταλήξουν στο 10. Καλωσορίζουμε επίσης το γεγονός ότι η κυρία Φερνιό με ιδιαίτερα ευνοϊκό τρόπο αντιμετωπίζει το θέμα του να γίνει κάτι για τους καταρτιζόμενους, τους υπομαθητεία βρισκόμενους. Αυτό είναι μια νέα προσέγγιση. Πρέπει να συνεισφέρουμε με περαιτέρω πληροφορίες εφόλων αυτών. Αλλά εδώ επικεντρωνόμαστε στους νέους που, αντιδρούν, που αντιμετωπίζουν ανεργία στην Ευρώπη και πρέπει να βρουν κάποια πορεία στο μέλλον. Ε, εδώ πρέπει να τους βοηθήσουμε να βρούνε μια τέτοια δυνατότητα δυνατότητα. Καλό θα είναι αυτό για την κινητικότητα των νέων και την απασχόλησή του στην Ευρώπη. Επίσης, ε, ε, τέθηκε ένα άλλο ερώτημα. Θέλω να υπενθυμίσω το θέμα τη μοναδική θηρίδα είναι για να μπορεί κανεί να αποστέλει, να αποστέλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και από αυτή τη θηρίδα να λαμβάνει την απάντηση. Σε σχέση με τα κράτη-μέλη λοιπόν, αυτό είναι το, εκείνο το οποίο διευκολύνει. Αν έχει κανείς ε, τα επαγγελματικά προσόντα και θέλει να στραφεί σε κάποιον να αποσαφηνίσει κάποια θέματα, Υπάρχει υφιστάμενη δομή, εμείς δεν προτείνουμε κάτι το διαφορετικό ή καινούριο. Τώρα σέθω στα διαφορετικά επαγγέλματα. Στο τέλος θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί και γιατί θέλουμε να εξευρεθεί μια λύση. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν κάποιες υπερβολές μεταξύ των μεν και των δε σε σχέση με κάποια επαγγέλματα. Από την άλλη πλευρά έχουμε και την ομολογία του ΔΕΚ και πρέπει να βρούμε τη χρυσή μέση οδό ε, για να προχωρήσουμε, για να μην ε, δημιουργηθούν προβλήματα. Πρέπει να τα εξετάσουμε αυτά σε μεγαλύτερο βάθος όσον αφορά τις επιπτώσεις, repercussions. Να δούμε πώς θα εξευρεθεί μια βιώσιμη λύση, αξιόπιστη λύση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά. Αυτόματη αναγνώριση τώρα και τροπολογία υπαριθμών 75. Αυτό είναι πραγματικά σοβαρή υπόθεση για μας και όσον αφορά την ε, προτεραιότητα υπό την, ε, το νομικό πλαίσιο για την εσωτερική αγορά, θέλουμε όλοι να είμαστε υπέρ η αυξημένη κινητικότητα. Η αυτόματη λοιπόν αναγνώριση είναι ένα μέσο να διευκολύνουμε την κινητικότητα. Αν θέλουμε να περιπλέξουμε τα θέματα τη αυτόματη αναγνώριση, αυτό είναι εκείνο το οποίο επιθυμούμε. Όσον αφορά το αρχικό πλαίσιο συζητήσεων για την προαγωγή τη ενιαία εσωτερική αγορά, α το ξαναδούμε λοιπόν αυτό παρακαλώ. Η αυτόματη αναγνώριση είναι κάτι για το οποίο δίνεται αγώνας, μάχη επί δεκαετίες και νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν θετικό. Τέλος, εξίσου σημαντικό όμως, οι αδερφές νοσοκόμες. Και να μην ξεχνάμε και τις ΜΕΕΣ βέβαια. Ανάφεραν πολύ, ανέφεραν πολύ τις ε, νοσοκόμες, αλλά εδώ εμπλέκονται και οι ΜΕΕΣ. 12 χρόνια, 12 χρόνια σχολικής εκπαίδευσης. Αν λαμβάναμε υπόψη και τον υπηαγωγείο θα καταλήγαμε με νοσοκόμες 16 ε, ή 17 ετών ηλικίας και κανείς δεν θέλει νοσοκόμες τόσο νέες να εργάζονται με πλήρεις ευθύνες στα νοσοκομεία. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και είμαστε διατεθειμένοι να εξευρεθούν, να βρούμε συμβαστικές λύσεις και θέλουμε και πάλι να συνεισφέρουμε και εμείς για την εξέβρεση συμβασμών και λύσεων. Στο τέλος πρέπει να εξευρεθούν συμβιβασμοί, συμβαστικές λύσεις. Η τελευταία μου παρατήρηση, αν ναι, είχαμε μετά και Πολωνέζες νοσοκόμες και Ρουμάνες νοσοκόμες. Σωστό. Ο κύριος Μπουσόη το έθιξε νομίζω αυτό. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν εμπεριέχονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προαναγγείλαμε μια αξιολόγηση στην δική μας πρόταση σε σχέση με αυτά. Ακόμα δεν έχουμε υιοθετήσει μια τελική θέση επ' αυτών. Ας αναφέρω δύο στοιχεία σε σχέση με αυτά για τις Πολωνέζες νοσοκόμες. Είναι μια συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών και της Πολωνίας ε, που κρατάει πολλά χρόνια. Έχουμε πείρα που έχει, έχουμε συλλέξει, ε, έχουμε συσσωρεύσει, πολλές συζητήσεις έγιναν. Και η Πολωνία το 2004 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάτι το, από το 2015-2016 θα ίσχυε. Έχουν προχωρήσει πολύ έχουν προχωρήσει. Για τις Ρουμάνες νοσοκόμες ακούσαμε πολύ προσεκτικά τα επιχειρήματα. Είναι όμως μια νέα, νεότερη, καινούρια κατάσταση. Εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιστερότερα η Ρουμανία και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει αυτό να προχωρήσει σε σχέση με την αυτόματη αναγνώριση. Να μην αφαιρεθούν δυνατότητες ελέγχων από τα κράτη υποδοχής, για παράδειγμα. Αυτά θα ήθελα να πω όσον αφορά το επάγγελμα των νοσοκόμων. Ας ολοκληρώσουμε τους φαρμακοποιούς. Θα θέλαμε προσεκτικά να εξεταστούν οι προτάσει τη κυρία Βερνιό για την επέκταση των δραστηριοτήτων των φαρμακοποιών, να δούμε αν αυτό είναι αναγκαίο ή όχι ως στοιχείο. Το έχουμε υπό εξέταση, δεν έχουμε ακόμα τελεσίδικα τοποθετηθεί. Μια ερώτηση επιπλέον, γιατί προτείνει η οχι ω στοιχειο το εχουμε υπο δεν εχουμε ακομα Επιτροπή την διαγραφή του άρθρου 21 εδαφίου 4 για την, το άνοιγμα νέων ε, φαρμακείων. Έχουμε κάποια κράτη-μέλη που έχουν σημαντικά επιχειρήματα εναντίον. Ανεκδοτολογικά να σας πω, σε σχέση με την Επιτροπή Αναφορών, γιατί ένας Γάλλος δεν θα μπορούσε να ανοίξει φαρμακείο στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλαξαν τα πράγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, άλλαξε το θέμα της εξαίρεσης. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία συζητούμε εδώ. Είναι μια αγορά που θέτει συγκεκριμένες δυσκολίες ε, για αυτό το επάγγελμα. Ίσως ε, ελπίζουμε όμως ότι μπορούν να εξευρεθούν και καλές ε, προτάσεις να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Συνοψίζω, πιστεύω ότι ακολουθεί μια κατεύθυνση αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή που πραγματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε τα όσα γίνονται από εσά όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω στην εισηγήτρια πλέον. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Βερνιό. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και πριν από τους συντονιστές έχουμε και άλλη συζήτηση. Λοιπόν, εγώ σημείωσα προσεκτικά όλες τις σκέψεις που ακούστηκαν, όπως και την προηγούμενη φορά σήμερα. θα ήθελα να πω ότι η επαγγελματική κάρτα, η επαγγελματική ταυτότητα είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο όχι μόνο για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελματιών όταν κυκλοφορούν, η κινητικότητά τους είναι πλέον απαραίτητη για τους νέους για να μπορέσουν να βρουν ένα επαγγελματικό μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο λοιπόν και θα συμφωνήσουμε όλοι. Θα ήθελα να υποστηρίξω επίσης την Επιτροπή όταν αναφέρεται στο θέμα της αυτόματης αναγνώρισης. Είναι αλήθεια ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα στους επαγγελματίες και στα κράτη-μέλη αυτή η επαγγελματική αναγνώριση αλλά είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να το έχουμε πάντα μπροστά μας, γιατί η κινητικότητα στην παρούσα φάση δεν είναι σημαντική τόσο πολύ, αλλά θα γίνει πολύ πιο σημαντική τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας για να διευκολύνουμε τη λεγόμενη θετική κινητικότητα και για τους επαγγελματίες και για το σύνολο των πολιτών. Ένα λοιπόν θέμα είναι η πολιτική, η γραμμή την οποία ακολουθούμε σε σχέση με, τα ευαίσθητα, με τις ευαίσθητες πλευρές, η διτή μορφή της κατάρτισης, ο χρόνος που απαιτείται για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες φάσεις. Είναι σαφές ότι η οδηγία αυτή δεν θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ βιαστικά, εάν υπάρχουν πάρα πολλές ε, αμφιβολίες. Θα πρέπει να υπάρξει μια σαφής ε, διαφανή εικόνα για το σύνολο των ε, πολιτών και για τις αρμόδιες αρχές, είτε θα έλεγα περιφερειακές, είτε εθνικές, δεν, είτε επαγγελματικέ, δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον Ευρωπαίο πολίτη να νιώσει ακόμα πιο Ευρωπαίος. Η συνεργασία ανάμεσα λοιπόν στα θεσμικά όργανα και τις πολιτικές ομάδες συνεχίζεται. Ευχαριστώ. Πράγματι εφόσον μπορέσουμε να καταλήξουμε και στον τομέα της εκπαίδευσης και στα ελάχιστα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα. Λοιπόν, κλείνουμε με το σημείο 10, περνάμε στο σημείο 11. Να πω για το 10 ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 15η Οκτωβρίου και θα εξεταστούν οι τροπολογίες στις 6 Νοεμβρίου Προθεσμία για κατάθεση συμβιβαστικών 27 Νοεμβρίου. Περνάμε τώρα στο 11. Ε, γνωμοδότηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κοφεράτη. Παρακαλώ, να μην κάνετε θόρυβο για να ακούσουμε τα σχόλια του εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν από οτιδήποτε άλλο τους σκιώδεις εισηγητές και τους συναδέλφους οι οποίοι πήραν μέρος ε, άμεσα στη συζήτηση που προηγήθηκε και το κάνω αυτό όχι τυπικά, όχι γιατί συνηθίζεται αυτό, αλλά το κάνω γιατί θεωρώ ότι υπήρξε πράγματι σημαντική επιθυμία για συμμετοχή των συναδέλφων πάνω στα δύσκολα σημεία, τα οποία μέσω της συζήτησης θα μπορέσουμε να λύσουμε, να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις οι οποίες ε, θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν θέσεις που πολλές φορές είναι η μία μακράν της άλλης. Όπως είχα ήδη πει, πάνω σε συγκεκριμένα θέματα όπως το θέμα της προώθησης των αυτοκινητοδρόμων της θάλασσας, των αερολιμένων, των χρηματοδοτήσεων, των μεταφορών, έχουμε βρει κάποιες λύσεις οι οποίες είναι θετικές. Έχουν μείνει βέβαια σε εκραμότητα και έχουν, ε, θα έλεγα, προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις και όχι αδικαιολόγητα. Τέσσερις, ε, τέσσερα σημεία πάνω στα οποία νομίζω έχουμε να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Αναφέρομαι στους συναδέλφους οι οποίοι δεν πήραν μέρος στην τελευταία φάση της συζήτησης που έχουμε κάνει. Θα ήθελα να τους ενημερώσω για τις συμβιβαστικές προσπάθειες που έχουν γίνει πέραν αυτού σχετικά με τις προθεσμίες. Έχουμε νομίζω ε, σεβαστεί τις προθεσμίες τις οποίες προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπουμε την δυνατότητα αναθεώρησης στα πλαίσια της ε, ρύθμισης που προβλέπεται στον κανονισμό στο άρθρο 57 έτσι ώστε να μην στερήσουμε την δυνατότητα περαιτέρω σε ένα κράτος μέλος να μπορέσει το συγκεκριμένο να, ε, να έχει στη διάθεσή του τις ίδιες δυνατότητες με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Στα θέματα της διακυβέρνησης, η τροπολογία της συναδέλφου Ιβάνοβα μας επέτρεψε να ορίσουμε ε, με ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο τα κράτη-μέλη μαζί με τον συντονιστή και σε συνεργασία με την πλατφόρμα για τους διαδρόμους θα προετοιμάσουν ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου διαδρόμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιτρέψει να συνδυάσουμε, όπως είπα, απόψεις οι οποίες αρχικά ήταν μακράν η μία της άλλης. Έχει σημασία εδώ και το σημειώνουμε στην αιτιολογική σκέψη και όχι στο κείμενο γιατί δεν είναι άμεσα σχετικό με τη γνωμοδέτησή μας, αλλά έπρεπε να το υπογραμμίσουμε ε, να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τους επιβάτες. Τέλος, νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε και για τους εσωτερικούς, ε, ε, εσωτερικές οδούς ναυσιπλογίες. έτσι ώστε να δώσουμε εγγυήσεις σε μια συγκεκριμένη πρόταση εάν εν καιρό βελτιώσει τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, να μπορέσει να επανεξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη σύνδεσή του με το δίκτυο, ε, στην ουσία δηλαδή να προβλέψουμε την λύση την οποία έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει για το σύνολο των TNTs. Νομίζω λοιπόν ότι για αυτούς τους λόγους τους οποίους ε, σας παρουσίασα έχουμε συνολικά μια καλή ισορροπία η οποία ανταποκρίνεται στην αρχική μας ιδέα που έχει σχέση την ενίσχυση, ε, την ενιοποίηση της μορφής του δικτύου και την θετική σχέση που πρέπει να έχει το δίκτυο με τους χρήστες από τη μία, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν δυσκολίες και με το περιβάλλον από την άλλη. Μιλάμε για διαρθρωτικές παρεμβάσεις οι οποίες δεν θα συμβούν μόνο σε ένα πράσινο χωράφι, αλλά για δίκτυα τα οποία εδώ και αρκετό καιρό λειτουργούν, μέσα στα οποία ζουν κοινότητες που έχουν αναπτύξει συνήθειες, ήθη θα έλεγα, και ακριβώς από εκεί έλκουν τα χαρακτηριστικά τους, την ταυτότητά τους. Λοιπόν, με όλα αυτά τα στοιχεία μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα των TNTs, όχι μόνο να προωθήσουμε τον αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα σε διαφορετικά δίκτυα, αλλά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συνδυασμό τους, να μειώσουμε το περιβάλλον, να σεβαστούμε ε, τα δικαιώματα των πολιτών και των μεμονωμένων και τα συλλογικά τους δικαιώματα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ρυθμίσεις, επιμέρους ρυθμίσεις ή εντάξει στο αρχικό πλαίσιο, ε, στο οποίο αρχικό πλαίσιο πολλά προσπαθήσαμε να προβλέψουμε, αλλά όχι φυσικά τα πάντα. Έτσι λοιπόν, η διαδικασία που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα φάνηκε ότι βοηθάει. Είμαι ικανοποιημένος λοιπόν στην ε, εργασία στην οποία καταλήξαμε. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα σχολιάσουν οι σκιώδεις και οι συνάδελφοι ε, μέλη της Επιτροπής που έχουν καταθέσει τροπολογίες. Ευχαριστώ Σέρτζιο. Oh, it is... Η κυρία Ιβάνοβα, όχι, ο κύριος Βάμπ πρώτα. Ούτε η παρακαθήμενη είναι η κυρία Ιβάνοβα, ούτε εγώ είμαι η κυρία Ιβάνοβα, αλλά την αναπληρώνω. Ε, λυπούμε που έλαβα το λόγο πολλές φορές σήμερα. Θα ήθελα πάντως να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κομφεράτη για το πραγματικά πολύ αξιόλογο έργο του στο θέμα αυτό και εκ μέρους της κυρίας Ιβάνοβα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που με τις τροπολογίες τους συνέβαλαν στη βελτίωση ε, του κανονισμού. Ήταν πολύ επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή και αυτό αποτυπώθηκε σε μια σειρά συμβαστικών τροπολογιών που λαμβάνει υπόψη και τις θέσεις του ΕΛΚ. Γενικώ δεν υπήρχαν αντιφατικά ή επίμαχα σημεία στις συμβαστικές τροπολογίες. Ένα ήταν μόνο το επίμαχο θέμα. Αφορά τη συμβαστική τροπολογία 10 που προβλέπει ότι αποδεικνύει σαφή προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία από οικονομική, οικολογική και περιβαλλοντική ε, προοπτική. Δεν ξέρω αν επιμένει η και καλά η ομάδα των πρασίνων για την διατύπωση αυτή. Κατά τη γνώμη μου είναι άνευ ε, ουσίας και η κυρία Ιβάνοβα προτείνει να καταψηφίσουμε αυτή την προσθήκη. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά την ελαστικότητα για τις διορίες με βάση τις αξιολογίες που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκτιμηθεί η πορεία των προγραμμάτων και ίσως αναθεωρηθεί το χρονοδιάγραμμά τους. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ισορροπημένο. Επίσης, προσθέσαμε και την διαδικασία για να κερδίσουν το χαμένο έδαφος ε, οι νέες χώρες μέλη. Αυτό ήταν ένα αίτημα και της κυρίας Ιβάνοβα και της κυρίας Χάντζλικ, ε, της Πολωνής συναδέλφου συμφωνούμε ε, για την προ... περίληψη στο κείμενο την, ε, τη συμπερίληψη της ε, πλατφόρμας για τους επιβάτες προκειμένου να, εξασ... να εξασφαλιστεί καλύτερη ενημέρωση στους πελάτες, στάνταρ έκδοση εισιτηρίων και γενικώ τέτοια θέματα. Ευχαριστώ. Περιμένω και τις απόψεις των υπόλοιπων σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ομοιότητά σου με την κυρία Ιβάνοβα. Είστε φτιστοί και οι δύο. Ο κύριος Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και τα συγχαρητήριά μου προς τον κύριο Κομφεράτη. Είχαμε συνεργαστεί και στην Επιτροπή για την... της κρίσης. Ήταν πολύ αγαστή συνεργασία, παρόλο που η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί. Εν πάση περιπτώσει, έχω και εγώ κάποια σχόλια. Πιστεύω και εγώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν από κάποια χρονοδιαγράμματα και κάποιες προθεσμίες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ είμαι υπέρ της ευελιξίας και της ελαστικότητας αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι στις μέρες μας είναι κατάλληλη μέθοδος αυτή της ευελιξίας. Πολύ φοβάμαι ότι έτσι απλώς θα παραταθεί η διαδικασία. Έχω κάποιες επιφυλάξεις λοιπόν για την ευελιξία που προτείνεται όσο αφορά τις προθεσμίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, ούτε και αυτά είναι υποχρεωτικά για τα κράτη-μέλη. Υπάρχει δυνατότητα. Και εκεί είχαμε κάποιες διαφωνίες αλλά μπορώ να συμφωνήσω με το αποτέλεσμα τελικά. Πάντως η σαφής ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι η κατευθυντήρια γραμμή για την εφαρμογή ενό δικτύου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την έμφαση που δίνουμε στις αεροκατοικημένες περιοχές, νησιά, ορεινές ζώνες κτλ. Αλλά στόχος των δικτύων είναι να μειωθεί η συμφόρηση, η στενοπή, κυρίως ε, και να βελτιωθεί η καλύτερη διασύνδεση των κόμβων. Αυτός νομίζω ότι είναι ο πρωταρχικός στόχος του δικτύου. Και άλλωστε η συμπερίληψη των υποδομών στο δίκτυο γίνεται σε αρκετά μεταγενέστερη φάση της διαδικασίας. Λίγο καθυστερημένα κατά τη γνώμη μου. Καλή η προσπάθεια του εισηγητού, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις συμβαστικές τροπολογίες 16 και 17. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτή η συμφωνία. Ίσως εγώ δεν έχω τόσο δραστήριους ε, συναδέλφους από τον κύριο Σβάπ. Θέλουμε τα δίκτυα να είναι λειτουργικά όχι μόνο για την ε, διακίνηση των αγαθών και προϊόντων, αλλά και για την ε, κυκλοφορία των επιβατών και συμφωνώ με κάποιους τυποποιημένους τρόπους ταξιδιού στην Ευρώπη. Είμαι γενικώ υπέρ αυτής της ε, τυποποίησης. Αυτά. Η αμφιβολίες μου είναι μάλλον ίσονος σημασίας. Πολλές φορές πάντως η διαδικασία που εφαρμόζουμε στις επιτροπές μας είναι η προσθήκη στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μερικές φορές προτιμώ ε, αντί να προσθέτουμε, να αφαιρούμε κάποια σημεία από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Κύριε Ρίλα, ε, για τους πράσινου. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία με τον εισηγητή. Η θέση μου πάντα όταν πρόκειται για μια γνωμοδότηση, και εδώ έχουμε γνωμοδότηση, δεν είμαστε εμεί η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, να περιοριζόμαστε επί των δικών μα αρμοδιοτήτων και την συζήτηση την βρήκα κάπως παρεκκλίνουσα πρέπει να πω, διότι δεν είναι υποχρεωτικά τώρα η αρμοδιότητα της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αυτής. Και θέλω να δώσω δίκαιο στον Όλε Σμιτ σε αυτά που είπε δεν θα πρέπει κατά πρώτη γραμμή να θεωρούμε ότι είναι δική μας αρμοδιότητα σε σχέση με τις αραιοκατοικημένες περιοχές εμείς να δούμε τι πρέπει να γίνει. Εμείς ως Επιτροπή Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς δεν έχουμε καμιά σχέση όσον αφορά την άμεση αρμοδιότητά μας με αυτό. Θέλω να υποστηρίξω από πλευρά του εισηγητή την προσπάθεια προβληματίστηκε να δει πώς μπορούμε εμείς ξεχωριστά να συνεισφέρουμε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή για αυτό το θέμα. Καλό είναι ότι επιμένει και εμένει εδώ να υπάρξει ένα, να ασκηθεί πίεση για να προχωρήσει. Καλό είναι αυτό, αλλά κύριε Σουβάμπ, εσείς σε αυτό το οποίο υπενηχθήκατε και επειδή επί σύντομο διάστημα δεν πρόσεχα, δεν παρακολουθούσα τι είπατε, αν εννοείται το θέμα των συντονιστών και τον ρόλο των συντονιστών, είναι μια συνεισφορά που μπορεί να δώσει ξεχωριστά η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και ακολουθώ τον εισηγητή σε αυτό. Και τώρα αν βλέπετε κάποιες ελλείψεις πρέπει να μας πείτε περί τίνος πρόκειται, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορείτε να σχολιάσετε εσείς σύντομα κύριε Σβάμπ. Πρόεδρε, να αποσαφηνήσω. είναι πραγματικά σημαντικό για μένα να ξέρω αν η κυρία Ρούιλε και οι πράσινοι θέλουν να υποστηρίξουν το συμβαστικό κείμενο λέγοντας ότι και θέλουμε να καταδείξουμε ότι θα υπάρξει πρόσθετη ευρωπαϊκή αξία από το της μία φιλοπεριβαλλοντική, ε, φιλική προς την ε, κοινωνική πολιτική προσέγγιση. Αυτό ήταν το θέμα. Ευχαριστώ. Uh, then, Πρόεδρος, εντάξει, τότε προχωρούμε. Εσείς έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πιστεύω ότι η γνωμοδότηση είναι ισορροπημένη και λύθη υπόψη και η κατάσταση στις νέες χώρες μέλη έγιναν δεκτέ οι τροπολογίε και των Πολωνών αλλά και τη κυρία Ιβάνοβα. Επίση, πρόταση για μείωση του διοικητικού κόστου και ιδιαίτερε επιπτώσει στην οικονομία. Η ομάδα μου θα υπερψηφίσει τι περισσότερε τροπολογίε και τι συμβαστικέ τροπολογίε του εισηγητού και θεωρώ το πιο σημαντικό είναι η γνωμοδότηση να περιλάβει κάποιες εξασφαλίσεις για το διάλογο ε, μεταξύ πολιτών, τοπικών και εθνικών αρχών για την υλοποίηση των στόχων και των προγραμμάτων. Πιστεύω ότι ε, θα διαλυθούν οι φόβοι που έχουμε. Μιλήσαμε κυρίως για τις τροπολογίες 4, 10 και 18. Ε, οι συμβαστικές τροπολογίες 4 και 18 δημιουργούν κάποια προβλήματα. Μπορεί να υπάρχουν θετικά σημεία, αλλά νομίζω ότι θα είναι δύσκολο για τις χώρες που αντιμετωπίζουν κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Με εξαίρεση λοιπόν αυτές τις ε, δύο τροπολογίες, ε, συμφωνούμε με τη γνωμοδότηση του κ. Κοφεράτη και το συγχαίρουμε. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να είναι παρόν άλλος και ο Ούτε ζήτησε άλλο μέλος της Επιτροπής μας το λόγο. Οπότε θα ήθελα να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και να δώσω το λόγο στον κύριο Βάιτερς από τη Γενική Διεύθυνση MOVE. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον εισηγητή τη γνωμοδότηση και να τον συγχαρώ καθώ και τα μέλη τη Επιτροπή για το εξαιρετικό του έργο. Οι συμβαστικέ τροπολογίε είναι πολύ καλέ, μπορούμε να τι δεχτούμε και είναι απόδειξη τη εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με τον εισηγητή. Χαίρομαι και για την ε, συμφωνία που επιτύχαμε για τις, ε, για τις ε, προθεσμίες. Το ίδιο ισχύει και για τις τροπολογίες που μιλάει για την επαφή κρατών μελών και με το συντονιστή για τους διαδρόμους. Και εδώ ήταν εξαιρετική συνεργασία. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 10 που επισημάνθηκε ξεχωριστά, δεν έχουμε πρόβλημα με το κείμενο τη τροπολογίας αυτή. Ούτω ή άλλω, όταν γίνεται ανάλυση κόστου ωφέλου ε, ενό προγράμματο, λαμβάνεται υπόψη και η κοινωνική, οικολογική και η περιβαλλοντική διάσταση. Ε, πέραν της ανάλυσης κόστους ωφέλους. Το κείμενο τη τροπολογία 10 δεν μα ε, προβληματίζει, δεν μα ενθουσιάζει κιόλα. Κατά τη γνώμη μα είναι περιττή διατύπωση, θα μπορούσε κάλλιστα να διαγραφεί, αλλά δεν μα ε, δημιουργεί πρόβλημα ούτω ή άλλως. Ευχαριστώ τον κύριο Κοφεράτη και τα μέλη της Επιτροπής για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και σίγουρα μερικέ από τις τροπολογίε θα τις διαβάσω απευθείας στην Γενική Διεύθυνση Τραν για να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ και εγώ συγχαίρω τον εισηγητή μας τον κύριο Κοφεράτη και τους και για την αγαστή του συνεργασία. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο, 11 Οκτωβρίου. Αλλά ας ξαναδώσω το λόγο και πάλι στο συντάκτη γνωμοστέ. Κύριε Κοφεράτη, έχετε το λόγο. Ένα πράγμα θα πω μόνο. Καταρχάς σημείωσα τις παρατηρήσεις, ε, θα λάβω υπόψη μου τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Εν πολλής νομίζω τις είχα προβλέψει Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έκανε όλε Σμιτ σχετικά με την τάση που έχουμε να να αυξάνουμε το μέγεθος των κειμένων και όχι να προσπαθούμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα και συνοπτικά. Επί της ουσίας τώρα. Η τροπολογία βέβαια δεν είναι της κυρίας Ρούλε, ε, είναι της Γκουε και γι' αυτό ακριβώς δεν υπήρξε αντίδραση. Εγώ δεν θέλω να πείσω κανέναν, αλλά τέτοιες απόψεις όπως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι λίγο γενικές. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι προσπαθώντας μέσω της προσθήκης μας να καταστήσουμε πιο λειτουργική την προσπάθειά μας, να ξεκαθαρίσουμε την προστιθέμενη αξία την οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε. Το θέμα είναι να καταστήσουμε πιο ε, αποδοτικά τα δίκτυα για να βοηθήσουν και το οικονομικό και το κοινωνικό σύστημα, αν θέλετε. Εμείς ε, θέλουμε να μην αλλάξουμε το νόημα της πρότασης της Επιτροπής με το οποίο συμφωνούμε. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να αλλάξουμε το κείμενο, απλά θέλουμε το κείμενο να το αλλάξουμε όχι ως προς την ουσία του, αλλά να το καταστήσουμε πιο ξεκάθαρο και κατανοητό. Ευχαριστώ κύριε Κοφεράτη. Λοιπόν, τελειώσαμε με το 11. Ήταν το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Κλείνει η συνεδρίαση της Επιτροπής εδώ. Η επόμενη συνάντηση είναι αύριο στις 9 το πρωί. Και τώρα θα περάσουμε στη συνάντηση των συντονιστών. Θα ζητήσω από τον Μάλκολ να αναλάβει την Προεδρία.